Okay, let's start. Good to see you back in the hemicycle. Λοιπόν, ας ξαναρχίσουμε. Αν πω η αλληλεγγύη, ο θελοντισμός, ε, η βοήθεια για αλλαγή σε μια κοινότητα, είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά σημαίνουν πολλά για σας. Καλώς και πάλι στο ημικύκλο, στην καρδιά του Ευρωβουλής, για μια ιδιαίτερη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Μια νέα συναρπαστική πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Ναύρατζης, που είναι δεύτερη φορά σήμερα μαζί μας, ε, που φιλοξενεί αυτή τη συζήτηση. Θυμίζω στους ακροτάσμους μα ότι είστε υπεύθυνο για την παιδεία, την νεότητα και τον αθλητισμό και θα μας πείτε γιατί θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό το σώμα αλληλεγγύης. Τα επόμενα 90 λεπτά θα ανακαλύψουμε περισσότερα για αυτή τη νέα πρωτοβουλία και πιστεύω πως μέχρι να φύγετε από αυτήν την αίθουσα θα τα ξέρετε όλα για αυτό το νέο είδος εθελοντισμού και βασιζόμαστε σε εσά να το διαδώσετε και να πείτε και στους γύρω σας ε, περί τίνος πρόκειται. Και αυτό που κάνουμε με τα κοινωνικά δίκτυα σήμερα είναι λίγα. Γι' αυτό και έχουμε καλέσει δύο πολύ σημαντικούς bloggers με μεγάλη επιρροή που θα μας δώσουν ίσως κάποιες πληροφορίες ή θα μοιραστούν μαζί μας κάποια μυστικά για το τι να κάνουμε ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα σε αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία. Και φυσικά οι πρωταγωνιστές ε, αυτής της πρωτοβουλίας, οι ενώσεις, ε, οι εθελοντές ε, και οι δικαιούχοι βέβαια θα μας πούν πώς λειτουργεί. Αυτό το η Να αναμεταδίδεται στο website της εβδομάδας ε, της νεότητας ε, στο European Youth EU και θέλουμε όσο γίνεται περισσότερο να συμμετέχετε. Είναι μια συζήτηση. Παρακαλώ να χρησιμοποιήσετε λοιπόν το Twitter σας για να μας στέλνετε σχόλια, αντιδράσεις. Έχουμε δύο hashtag, τα βλέπετε εκεί στην οθόνη hashtag ε, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Βλέπετε εκεί στην οθόνη την ε, ορθογραφία και Youth Week. Και εγώ θα χρησιμοποιήσω το τηλέφωνό μου για να θέσω τις ερωτήσεις σας στον Επίτροπο και στους ομιλητές μας. Πρώτα θα στραφώ στον Επίτροπο. Είστε αρμόδιος για την επαιδεία, τον πολιτισμό, την νεότητα και τον αθλητισμό. Εσείς ξεκινήσατε αυτή την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ε, είδατε να αναπτύσσετε στα δυόμιση χρόνια ύπαρξή του. Καταρχάς πείτε μου γιατί ε, ξεκινήσατε αυτή την πρωτοβουλία. Καλησπέρα σας. Ε, είμαι ιδιαίτερα ευτυχή ευτυχής που είμαι σήμερα εδώ για να μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Σώμα ε, Αλληλεγγύης. Ήταν μια ειδική, ε, ιδιαίτερη πρωτοβουλία στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Ξεκίνησε ως μια συλλογική προσπάθεια για να δείξουμε ένα αυτό παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και για να μπορέσουμε να αποδείξουμε την ύπαρξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής ταυτότητας στους Ευρωπαίους πολίτες. Γι' αυτό αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την πρωτοβουλία για τους νέους γιατί βασικά εσείς είστε οι πιο προσιλωμένοι υποστηριχτές της Ευρωπαϊκής ε, Λελεγγύης και πιστεύουμε πως αυτό το project μπορεί να σας ε, ε, καλύψει σε εσά τις προσπάθειές τον ενθουσιασμό σας προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης αλλά μπορείτε επίσης να δώσετε το παράδειγμα για τις πιο ηλικιωμένες γενιές ώστε να ανανεωθούν και να τους προσελκύσετε πάλι στο ευρωπαϊκό project. Γι' αυτό και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στόχο είχε να στηρίξει τοπικές κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη σε περιπτώσεις επίγουσας ανάγκης ή στα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, υγειονομικής περίθαλψης, σε διάφορους θεσμούς και ε, άλλους τομείς της ε, ζωής της κοινωνίας. Και έχει ε, συναντήσει μεγάλη επιτυχία. Έχουμε 124.000 ε, ετούντες ε, και καθημερινά αναπτύσσουμε περισσότερες ε, ε, δραστηριότητες. Ελπίζω λοιπόν πως και στο μέλλον θα γίνει ακόμα πιο μεγάλο και πιο επιτυχές το πρόγραμμα και ελπίζουμε που θα εμπνεύσει ακόμα περισσότερους εκείνους που μας παρακολουθούν online αλλά και όσους βρίσκονται σήμερα εδώ στο ημικύκλιο. Είναι δύσκολο να μπει κανεί στο σώμα αλληλεγγύης. Χρειάζεται ιδιαίτερες δεξιότητες και γνώσεις. Όχι καθόλου. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης βασικά είναι προσπάθεια αντιστοίχησης. Υπάρχει μια ανάγκη και υπάρχει ζήτηση και προσφορά. Αν θέλει κανείς να είναι εθελοντής και ε, γράφεται, λέει ποιες είναι οι δεξιότητές του, περιγράφει το κίνητρό του και μπορείτε να βρείτε ΜΚΟ ή οργανώσεις. Επιπλέον μπορείτε να συνομιλήσετε με τους ε, ομολόγους σας και να φτιάξετε και κοινό πρόγραμμα. Μάλιστα, μας δώσατε ήδη κάποια αριθμητικά στοιχεία. 125.000 νέοι έχουν ήδη ζητήσει να γίνουν μέλη του Σώματος Αλληλεγγύης και σχεδόν 15.000 ήδη έχουν ολοκληρώσει τις δραστηριότητε τους είτε αυτή τη στιγμή ε, δρούν επί τόπου. Πώς σας κάνει να αισθάνεστε η ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας. Είμαι πολύ ευτυχής, ε, απαντά ο Επίτροπος, αν δούμε τα στοιχεία είναι σαφές πως υπάρχουν κάποιες ε, ε, πολύ δραστήριες χώρες όπου οι νέοι ε, δραστηριοποιούνται και στηρίζουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και την ιδέα της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης όπως είναι η Ισπανία, η Ιταλία, επίσης η Ρουμανία είναι οι πιο δραστήριες αλλά να τονίσω και την Τουρκία, όπου οι νέοι από την Τουρκία είναι πολύ δραστηροί και υπάρχουν πολλά αιτήματα που έρχονται από την Τουρκία. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα και είμαι ευτυχής γι' αυτό, διότι μπορούμε να περιλάβουμε κόσμο πέρα και από τα σύνορα της Ένωσης. και να δώσουμε νόημα ε, για τους νέους που ζουν ε, πέρα από τα κράτη της Ένωσης. Να έχουν την αίσθηση ότι ανήκουν σε αυτή την κοινότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντική, πιο σημαντική αποστολή. Να φτιάξουμε μια συνεκτική και ελκυστική κοινότητα. Τώρα το ενδιαφέρον των νέων ε, για αυτά τα προγράμματα τι σημαίνει, για πείτε μας δύο λόγια για την νέα γενιά της Ευρώπης. Σημαίνει ότι είναι δραστήριοι και ενεργοί, είναι προσιλωμένοι όχι μόνο σε μια δημοκρατική κοινωνία, αλλά θέλουν να κάνουν κάτι προς όφελος ε, της κοινότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εθελοντές που δουλεύουν στα διάφορα μέρη πηγαίνουν εκεί για να ε, αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες, να βοηθήσουν, να κάνουν φίλους, να βοηθήσουν τις τοπικές κοινότητες και να συμβάλλουν στο κοινό ε, καλό όλων των Ευρωπαίων. Να ρωτήσω και για το μέλλον του σώματος αλληλεγγύης. Πώς θα αναπτυχθεί κατά τη γνώμη σας εσείς. Κάνατε μια φιλόδοξη πρόταση για το επόμενο ε, προϋπολογισμό της Ένωσης. Φαντάζεστε ότι θα γίνει τόσο ε, σημαντικό όσο το έρασμος. Ελπι, το ελπίζω γιατί μέχρι στιγμής ε, είχαμε μεγάλες επιτυχίες όπως και με το έρασμος. Ε, μπορούμε να και θα αυξήσουμε στο 1,25 δις ευρώ για το επόμενο πολιετές μας πλαίσιο δηλαδή σημαίνει αυτό 350.000 νέους ε, που καλύπτονται από αυτήν τη νέα ε, αύξηση του προγράμματος πιστεύω πως οι, οι προοπτικές είναι πολύ καλές αν κανείς μείνει δραστήριος και διατηρήσει τη ορμή και την ένταση των δραστηριοτήτων θα είμαστε τόσο επιτυχείς όπως όσο και με το έρασμος. Σας ευχαριστώ λοιπόν, μας δώσατε το ιστορικό και τώρα θα ξεκινήσουμε την συζήτηση με κάποιους από τους ανθρώπους που έχουν ωφεληθεί από αυτά τα προγράμματα. Απλά να σας θυμίσω πως έχετε τα ακουστικά που σας, με τα οποία ακούτε τις μεταφράσεις από 22 νομίζω γλώσσες λέει ο μιλητής. Μπορείτε να ακούσετε ε, λοιπόν ε, τη μετάφραση, στη διερμηνία. Να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τους διερμηνείς για τη σκληρή τους δουλειά σήμερα και θα ήθελα να περάσω στο πρώτο παράδειγμα όπου το σώμα αλληλεγγύης έκανε ε, τη διαφορά. Αναφέρατε την Όρτζια, ξέρετε τι συνέβη στην Όρτζια τον Οκτώβριο του 2016. Ένας ε, καταστροφικός σεισμός αυτή την πόλη της κεντρικής Ιταλίας άφησε πίσω του καταστροφή. Πολύ, πολλά κτίρια έπρεπε να ανοικοδομηθούν, Πολλοί κόσμοι χρήζονταν βοήθεια. Μια ομάδα του Ευρωπαϊκού Σώματο Αλληλεγγύη εστάλει εκεί για να προσπαθήσει μαζί με του υπόλοιπου. Δείτε λοιπόν τι έγινε. My name is Alexandra Maria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 Και πολλοί ακόμα εθελοντέ ε, πήγαν. Ακούσαμε την Άννα Μαρία από την Εστονία, τον Ροντρίγκο από την Πορτογαλία, τον Καν από την Γαλλία, μεταξύ άλλων. Και σήμερα θα σα παρουσιάσω αυτή την ιστορία τη Νόρτσα. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε εδώ μαζί τον Νικόλα Αλεμάνο, που είναι ο δήμαρχο τη Νόρτσα, ε, που ωφελήθηκε, πόλη που ωφελήθηκε από αυτή την προσπάθεια. Σα ευχαριστώ που ήρθατε στι Βρυξέλλε. Επίση είναι μαζί μα ο Τζόρτζ από την Ασοσιασιόν Εκόρα που είναι εκπρόσωπος της Ένωσης που κάνει διάφορα project στην Όρτζα One of the volunteers. Και έχουμε και έναν από τους εθελοντές, τον Τζακ, που ακόμα είναι στην Όρτζα Και τέλος υποσχέθηκα ότι έχουμε και online ε, ε, bloggers που θα μας δώσουν κάποια στοιχεία. Η Μπάσα Γραμπόσκα είναι blogger από το Gdansk ε, μια πόλη όπου η λέξη αλληλεγγύη σημαίνει πολλά. Θα ακούσετε λοιπόν την ιστορία, αλλά θέλω να ακούσω από εσά πώ μπορείτε να πουλήσετε αυτή την ιστορία στον κόσμο, γιατί θέλουμε ο κόσμο να μάθει περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Σώμα αλληλεγγύη. Να ακούσουμε τον Τζόρτζο από την Ένωση, τον Τζόρτζο από την Ένωση που για να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Έχουμε ένα τρίγωνο. Έχουμε έναν εκπρόσωπο της Ένωση, έχουμε έναν εθελοντή και έχουμε και τον ε, δικαιούχο. Πώς ήρθατε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη, πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας. Η οργάνωσή μας δεν έχει την έδρα της στην ε, Νόρτσα ακριβώς, το Τρασινιάνο είναι η έδρα μας και είμαστε πολλές ομάδες που ξεκινάμε από το Erasmus Συν. Ο σεισμός έγινε τον Αύγουστο και μετά έγινε και ένας δεύτερος τον Οκτώβριο. Τρεις ομάδες ε, είχαν χρηματοδοτηθεί από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα από εμάς. Τους ε, σεισμούς τους νιώσαμε και είδαμε και τι ειδήσει μαζί με του άλλου συμμετέχοντε την επόμενη μέρα και είχαμε αυτή την αίσθηση ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν είχαμε τα μέσα όμως. Ακόμα δεν είχαμε έρθει σε επαφή με τον Δήμαρχο και ευτυχώς μας προσκάλεσαν σε συνάντηση με τον Εθνικό Ιταλικό Φορέα και άλλες οργανώσεις από την περιοχή των, τη σεισμόπληκτη. Εκεί συναντήσαμε τον Νικόλα και αμέσως βρήκαμε έναν τρόπο να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Υποβάλαμε λοιπόν το project μέχρι τα τέλη Απριλίου και τον Αύγουστο στείλαμε τους πρώτους 16, ήρθαν οι πρώτοι 16 εθελοντές. Ε, στην Όρτσα είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανεί τι συμβαίνει. Πρέπει κανεί να πάει για να, να για να πει τι αισθάνεται. Την πρώτη φορά που πήγα, λοιπόν, φανταστείτε ότι είστε σε ένα μέρο που τα πάντα βρίσκονταν ε, μέσα στα τείχη μιας πόλης και ξαφνικά γίνεται ένας σεισμός και δεν έχετε δικαίωμα να περπατήσετε καν εκεί που περπατάγατε προηγουμένως στην καθημερινότητά σα. Ναι, είναι πολύ καλό που μας θυμίζετε το όλο πλαίσιο. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα για την πόλη τη Νόρτσα, αλλά οι εικόνε που βλέπαμε από την καταστροφή τότε ήταν πραγματικά συγκλονιστικέ. Εσεί, Δήμαρχε, όταν ακούσατε ότι υπάρχουν εθελοντέ από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε που ήταν έτοιμοι να έρθουν για να βοηθήσουν, τι σκεφτήκατε, τι ήταν το πρώτο που σκεφτήκατε. Θα μιλούσα αγγλικά στα όνειρά μου, αλλά εδώ προτιμώ να μιλήσω ιταλικά. Όταν τα παιδιά φτάσανε στην Όρτσα, η όλη κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Η πόλη είχε καταστραφεί και δεν είχαμε ούτε ένα μέρος ε, να τους προσφέρουμε στέγη. Ε, τα παιδιά κοιμήθηκαν εκεί που κοιμόμασταν κι εμείς, στις σκηνέ. Έφαγαν εκεί που τρώγαμε κι εμείς. Στις σκηνέ, κατά τις σκηνέ. Και επίσης έπρεπε να δουλέψουν όπως και εμείς στον δρόμο. Ε, συνάντησαν ανθρώπους που είχαν ανάγκη, η κοινότητά μας, οι κάτοικοι της Νότσα, είχαν ανάγκη να πάρουν ε, μια δόση θετικής ενέργειας. Τα παιδιά αυτά με την ζωτικότητά τους, με το κέφι τους, μπόρεσαν να το προσφέρουν με την διάθεσή τους να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ζήσαμε στιγμές σημαντικές, τρεις διαφορετικές εμπειρίες με τρεις διαφορετικές ομάδες και μια μελλοντική που θα έρθει τον Ιούλιο. Στην αρχή όλοι κάτοικοι, η κοινότητά μας έβλεπε με κάποια περιέργεια τα παιδιά αυτά τους νεαρούς που ακόμα και στους κρύους μήνες του χειμώνα κυκλοφορούσαν με ένα λευκό τισερτ που είχε πάνω τυπωμένο κάτι το, ένα έγχρωμο σύνθημα, ένα χρωματιστό σύνθημα. Μετά μπήκαν πραγματικά την καρδιά, στον πυρήνα τη κοινότητά μα ε, των κατοίκων μα και άρχισαν να έχουν ε, επικοινωνία και επαφή με του ηλικιωμένου, τους νέους, τα παιδιά. Με τα δικά μας τα παιδιά με ειδικέ ανάγκες. Και ήταν πραγματικά εντελώς στη διάθεσή μα θυμάμαι, πολύ καλά, αρκετέ σκηνέ. Με σημάδεψαν, θεωρώ, με τρόπο άκρο θετικό ε, με την παρουσία του μεταξύ των κατοίκων μα. Συμμετείχαν σε όλε τι κοινωνικέ μα δραστηριότητε. Και το 2017 θυμάμαι ότι όταν ε, μία Εστονή η Αλεξάνδρα που εμφανίστηκε στο βίντεο είχε πρόσβαση σε αυτήν την εκδήλωση ε, την ημέρα που ήταν και δική της εθνική γιορτή στο σχολείο ε, και δεν ε, μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της. Μετά θυμάμαι ότι παίζαν bridge νέοι με τους γέρους μας, ε, τους ηλικιωμένους μας, με ανθρώπους που δεν ήξεραν αγγλικά και προσπαθούσαν να του το εξηγήσουν με κάθε τρόπο, με τη γλώσσα του σώματος, με, με χειρονομίες ε, και να επικοινωνήσουν. Ή θυμάμαι τη δουλειά που έκαναν σε συνεργασία με τα παιδιά μας, πώς φτιάξαν πύληνα και κεραμικά για το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. Μιλάμε για μια πραγματική συμμετοχή στις παραδοσιακέ μα εκδηλώσει εκδηλώσεις με παραδοσιακές φορεσχές ε, στον επιτάφιο της Μεγάλης Παρασκευής που συμμετείχαν και φορώντας τα δικά μας, τι δικές μας στολές. Η παρουσία του στην κοινότητά μα προσπαθούσε να φέρει ε, αυτό που χρειαζόταν ε, στην κοινότητά μας, την κανονικότητα την ομαλή διεξαγωγή των γεγονότων. Τζακ, και εσύ από του εθελοντέ, μου αρχίζει πήγε σε μια συνέντευξη. Νομίζω την πρώτη φορά πήγε για δύο μήνε ε, στην Όρτσα, μετά πήγε πίσω στη Σουηδία για ένα μήνα και μετά ξαναπήγε στην Όρτσα. Το μέρο ε, τραβάγε κοντά του. Μπορείς να εξηγήσεις τι κάνεις σε καθημερινή βάση. Ποιος είναι ο ρόλος ως εθελοντή στην όρθα. Ε, το πρώτο είναι ότι συνεπάρχουμε με άλλους Ευρωπαίους εθελοντές. Όλοι είναι ενθουσιώδεις. Θέλουν το μέρος γύρω τους να γίνει καλύτερο. και δεν υπάρχει χειρότερο μέρο για να το κάνει κανεί αυτό από την Όρτσα αυτή τη στιγμή. Η ενέργεια που υπάρχει εκεί είναι πολύ σημαντική και μας βοηθάει. Σε καθημερινή βάση. Κάναμε πολλά θεατρικά εργαστήρια. Κάθε μέρα πηγαίναμε στο σχολείο και όπως είπε και ο Νικόλα, η συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις ήταν πολύ σημαντική Μάλιστα, έχετε δηλαδή πολύ αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα. Μιλάτε τελικά. Ε, πολύ καλά μιλάω. Και παρόλα αυτά καταφέρνετε να επικοινωνείτε με ηλικιωμένους, με όλους τους νέους που καταφέρνετε να βοηθήσετε. Ναι, το σημαντικό είναι να μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια γραμμή επικοινωνίας. Είναι θέμα θέλησης να θέλει κανείς να βοηθήσει. Έτσι γίνεται ε, ε η διασύνδεση. Άρα μας λέτε ότι η γλώσσα δεν είναι φραγμός. Ε, γι' αυτό το λέω για όσους μας ακούτε και σκέφτεστε... θα ήθελα να μπορώ να το κάνω, αλλά θα χανόμουν στη μετάφραση. Ναι, η γλώσσα μπορεί να είναι ένα φραγμός, αλλά μπορεί κανεί και να τον υπερβεί. Και αυτή η εμπειρία, πώ σα έχει αλλάξει ω άνθρωπο, αν σκεφτείτε όλο αυτόν τον καιρό που περάσατε στην Όρτσα, πώ σα άλλαξε ω Ευρωπαίο πολίτη κυρίω. Ε, το 2016 όταν ξεκίνησα μου φαίνονταν όλα αυτά πολύ μακρινά σαν να μην μπορούσα να κάνω τίποτα όταν όμως δίνει στον κόσμο μια ευκαιρία να κάνει κάτι για τα γεγονότα που συμβαίνουν ανά την Ευρώπη δεν κάνουν μόνο καλά αλλά αρχίζουν και νοιάζονται κιόλα για το τι συμβαίνει σε αυτή την ένωση. Αισθάνονται ότι του επηρεάζει ό,τι και αν συμβεί. Το όντι. Νομίζω ότι έτσι αισθάνεται κανεί όταν βρεθεί εκεί και βλέπει και τι ανάγκε τη τοπική κοινότητα. Επίση, μια τελευταία ερώτηση προ τον Τζο. Ξέρει τώρα τι μπορεί να κάνει το σώμα αλληλεγγύη για να βοηθήσει οργανώσει σαν τη δική σου. Τι θα πρέπει να αλλάξει να ξανασχεδιαστεί σωστά. Το πρόγραμμα είναι πολύ ευέλικτο. Ε, Επιτρέπει στους οργανισμούς που οργανώνουν, αυτούς που συντονίζουν, να βρουν την καλύτερη λύση. Η πραγματική επιτυχία για μας, ας πω, στο πρόγραμμα αυτό, είναι ότι καταφέραμε να συμφωνήσουμε αυτό το τρίγωνο συνεργασία που περιγράψατε. Εάν δεν είχαμε καλή συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, ο Επίτροπος είπε πάντρεμα Τέτοιο δεν έπρεπε να είναι. Ναι. Διότι, όπως είπα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα χωρίς τη βοήθειά τους. Παρομοίως και εκείνοι δεν θα μπορούσαν χωρίς εμάς. Και χωρίς τους εθελοντές θα μπορούσαμε να έχουμε υποβάλει ένα πολύ ωραίο project και να μην γίνει τίποτα. Να μείνει θεωρητικό. Νομίζω η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει κανείς όταν δουλεύει σε μια πληγήσα περιοχή είναι ότι είναι πολλά αυτά που έχει να κάνει. Οι εθελοντές μπορούν και αυτό μπορούν να προσφέρουν και οι Ευρωπαίοι είναι η κοινωνική διάσταση, η ανθρώπινη επαφή, να μιλάνε στους ανθρώπους, να νιώθουν ότι η Ευρώπη είναι κοντά τους και επίσης να δείχνουν και στην Ευρώπη τι συμβαίνει γύρω τους, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όπω είπε και ο Τζακ, έχει αλλάξει η στάση του. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει λίγη μεγαλύτερη συμμετοχή. Συμμετοχή στο κατασκευαστικό κομμάτι. Να βοηθάμε στην ανοικοδόμηση, στην εκκλησία, στην ε, απομάκρυνση των ε, ε, συντριμιών. Αλλά χρειάζονται πολλά μαθήματα ασφάλειας ε, που πρέπει κανείς να μάθει και να κάνει πριν μπορέσει να βοηθήσει. Γι' αυτό για μας είναι πολύ καλύτερο να βοηθάμε και να ενισχύουμε στην κοινωνική διάσταση. Οι δεξιότητε που χρειάζονται εκεί δεν είναι τόσο εξειδικευμένε. Μπορεί κανεί να πάει απευθεία και να αρχίσει να κάνει κάτι, να προσφέρει. Δεν χρειάζεται να είναι μηχανικό. Εντελώ. Και μπορεί επίση να το κάνει αυτό με πάθο. Ε, και Πέτρο Ναύρατσιτ, θα ήθελα να συμμετάσχετε κι εσεί, γιατί νομίζω το Σεπτέμβριο του 2017 επισκεφθήκατε την Όρτσα και δηλώσατε τότε ότι η Όρτσα είναι ένα υπόδειγμα ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Θα ήθελα να μου πείτε τι, πώς σας φαίνονται οι μαρτυρίες που ακούσαμε. Αυτό που είπε ο Τζον το πιο σημαντικό νομίζω. Η ανοικοδόμηση τις σεισμόπληκτες περιοχή, δεν απλώς ανοικοδόμηση των κτηρίων που έπεσαν και του υλικού περίγυρου και των κτηρίων αλλά είναι θέμα αποκατάστασης ψυχικής ε, οι κοινότητε αυτέ, οι κάτοικοι αυτοί που αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι, να αισθανθούν ότι περιβάλλονται από ανθρώπινη φροντίδα. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύη μπορεί να έχει και συμβολική αξία αλλά για την ε, ψυχολογική υποστήριξη του κόσμου είναι πρωταρχική σημασία σε βοήθεια. Είναι ένα μήνυμα από τον εξωτερικό κόσμο ότι τους χρειάζεται ακόμα και ότι όλοι παρακολουθούν το τους συμβαίνει, ότι όλοι τους ακούν, ότι όλοι θέλουν να τους βοηθήσουν. Είναι σημαντικός παράγοντας για την επιβίωση μιας κοινότητας και για την ενίσχυση τη καλή τη κατάσταση. Και μια τελευταία ερώτηση προ τον Δήμαρχο. Όταν επισκέφθηκε ο Δήμαρχο στην Ότσα, όταν έρχονται Ευρωπαίοι πολιτικοί και ηθήνοντες να επισκεφθούν και εθελοντέ. Για τους κατοίκους είναι ένα μήνυμα ότι δεν είναι μόνοι. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη φαίνεται να έχει κάποιο νόημα. Είναι έτσι. Κοιτάξτε, ε, πιστεύω ότι με το Σώμα Αλληλεγγύης και τα Ευρωπαϊκά Σώματα Αλληλεγγύης η Ευρώπη έχει έρθει πιο κοντά στους πολίτες της. Και αυτό μέσω των ε, πιο νέων κιόλας από τους πολίτες μας. Έχουν δείξει ότι υπάρχει ε, ουσία και υπάρχει και νόημα κάτι που μπορεί να κάνει όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς να αισθανθούν πιο κοντά μεταξύ τους και αυτό είναι αλληλεγγύη εμείς πραγματικά αισθανθήκαμε αυτή την οικειότητα, αυτή την εγκύτητα προς όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς μέσω των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που ήρθαν να μας επισκεφθούν. Ο Επίτροπος Ναυράξιξ ήρθε να μας επισκεφθεί, το ίδιο και αποστολή από το Κοινοβούλιο, Επίτροπος Κρετσού εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών αυτό έφερε πραγματικά ένα κύμα αισιοδοξία, ε, ιδίω από τους νεαρούς θελοντές και αυτό επέτρεψε στην πόλη μας να αισθανθεί ότι είναι κοντά της τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ότι είναι κοντά της οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι Αυτό πραγματικά κατέριψε υλικά όλους τους φραγμούς. Δεν θα άλλαζα πολλά σε όλο αυτό το πλαίσιο. Απλώς θα επέτρεπα σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους εθελοντέ, να μπορέσουν να παρατείνουν αυτού του είδους ε, την ε, εμπειρία. Τους είδα να φεύγουν από το χωριό μας, από την πόλη μας, με τα δάκρυα στα μάτια για να θέλουν να ξαναγυρίσουν. only one getting <laughs> applause. And please send us your reaction. Στείλτε μας τις αντιδράσεις σας στο Twitter. Εδώ είναι το hashtag Youth Week EU Solidarity Core. Θα είμαι πολύ περίεργος να μου πείτε τη γνώμη σας για όσα ακούσατε. Τώρα η Βάσα Γκραμπόφσκα είναι blogger και επηρεάστρια online Έχετε πολλούς follower. Σας παρακολουθούν πολύ καθημερινά. Θέλω λοιπόν να μας πείτε κι εσείς κάποιες ιδέες. Ακούσαμε μια ιστορία που είναι συγκινητική κιόλα για, για τους ανθρώπους, για μια κοινωνία και κοινότητα που πρέπει να νοικοδομηθεί. Ε, θα λέγατε και τη συχαίνω αυτή τη λέξη ότι θα πούλαγε αυτή η ιστορία καλά στο διαδίκτυο. Ασφαλώς, γιατί είναι πολύ συγκινητική, γιατί και εγώ, να σας πω, δάκρυσα. Δάκρυσα από αυτά που μας είπατε. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να διαδώσουμε αυτό το μήνυμα και πιστεύω ότι όλα στο διαδικτύο, το Instagram, το YouTube, τα blog έχουν να κάνουν με το συνέστημα. Αν κάποιος λοιπόν μπορεί να ανταποκριθεί στο περιεχόμενο που δημοσιεύεται, αυτό αποτελεί επιτυχία. Αυτό το project δηλαδή, λοιπόν, όλη η δουλειά αυτή που κάνατε, μπορεί να πουλήσει καλά και είναι ατυχές το ότι χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση γιατί είναι από άλλη σφαίρα αλλά πιστεύω ότι ναι, αποτελεί κάτι τέτοιο. Τι είδους ιστορία λοιπόν θα θεωρούσατε ότι θα ήταν ενδιαφέρουσα. Κάποιος σαν τον Τζακ θα ήταν ενδιαφέρον να τον παρακολουθείτε στην καθημερινή του δουλειά, στις συναντήσεις του με τους νέους τέτοιου είδους ιστορίες να έχουμε υπόψη μας γιατί θέλουμε να μάθει πιο πολλοί κόσμος τι κάνουν οι εθελοντές επιτόπου απάντηση νομίζω ότι θα πρέπει να παρουσιάσετε δύο πλευρές Έχουμε αυτό το τρίγωνο, όπως είπατε και προηγουμένως. Είναι σημαντικό λοιπόν να δείξουμε τις απόψεις ε, και των δύο πλευρών. Και αυτού που δίνει τη βοήθεια και αυτού που δέχεται τη βοήθεια. Το project σας ε, στο διαδικτυό με συνάρπασε. Γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί δίνετε καθημερινές, συγκινητικές ιστορίες που ε, έχουν να κάνουν με εσάς, τους εθελοντές και τους ανθρώπους που βοηθάτε. Θα πρέπει λοιπόν πάντα να έχουμε υπόψη μας αυτά τις δύο πτυχές του προβλήματος, του project μάλλον. Αυτό που μπορώ να σας πω σε ειδική σε τέτοια θέματα είναι το YouTube το οποίο αναφέρεται δεν έχετε, έχετε YouTube. Δεν σας έχω ακολουθήσει εκεί πέρα. Δεν έχουμε πολύ... Μάλλον ε, έχουμε πολύ περιεχόμενο, δεν έχουμε πολλά like. Ναι, αυτό το πρόβλημα το έχουμε. Αν μπορείτε να κάνετε like λοιπόν στη σελίδα μας. Η δουλειά σας είναι συναρπαστική και πολύ εκτενής. Και νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να τη γνωρίζει πιο πολλοί κόσμος. Να τους κάνετε λοιπόν like στην σελίδα του στο, στο facebook και να γίνετε συνδρομητές. Ε, μάλιστα. Τι είδους ιστορίες λοιπόν δημοσιεύετε online. Αυτό που κάνουμε συνήθως ε, στην Όρσια είναι να δίνουμε πρόσβαση σε έναν από τους αθλητές ε, στα social media. Μαζεύει τις ιστορίες λοιπόν από όλους και ο καθένας γράφει 500 ε, χαρακτήρες γιατί έρχονται και στο τέλος βάζουν άλλες 500 χαρακτήρες για το τι έκαναν και κάνουν συμφωνίες και με τους ε, ντόπιου. Έχουμε λοιπόν και τις δύο πλευρές, και τις εκ των και τα, εκ από τα έξω. Έχουμε και τους ε, μόνιμους ε, ε, που κάνουν μια εκπαίδευση στην αρχή και μετά και τα δικά τους στοιχεία μπαίνουν ε, online. Έχουμε λοιπόν ε, μία σελίδα για το VoloTube και μία σελίδα για τους θελοντές για την Όρτσια. Μάλιστα. Μα είπε, ε, Τζακ, ότι λαμβάνετε πολλά, μάλλον δεν δίνετε πολλά, αλλά λαμβάνετε και πολλά. Και μα είπατε πώ αυτή η εμπειρία άλλαξε τη ζωή σα. Και σύντομα θα επανέλθετε στη Σουηδία, στη Στοκόλμη. Τι θα κάνετε λοιπόν στη συνέχεια, θα συνεχίσετε να εργάζεστε ω εθελοντή. Τι έχετε υπόψη σα, ποια είναι τα σχέδιά σα. Πολύ καλή ερώτηση. Σίγουρα θα συνεχίσω να κάνω έργο για τη δική μου κοινωνία, κοινότητα. Δεν ξέρω που θα πάω βέβαια. Αλλά σίγουρα θα εργάζομαι για την κοινότητα. Γιατί υπάρχει πάντα μεγάλη, μεγάλη ανάγκη. Να βοηθάμε την ε, τοπική κοινωνία. Και ίσως ε, βρω και μία δουλειά, δεν ξέρω, θα δω. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για όλα αυτά που κάνατε. Και μια τελευταία κουβέντα προς τον Δήμαρχο. Η πόλη δεν έχει ακόμα ανοικοδομηθεί. Υπάρχουν ακόμα πολλές ελλείψεις και πολλές ανάγκες. Τι θα ελπίζατε λοιπόν να δείτε από την ε, νέα φρουνιά ε, αθρεντών στην Ορσία. 16 ναι, ε, θα υποδεχτούμε ακόμα 16 παιδιά στις, ε, τον Ιούλιο, τον επόμενο Ιούλιο. Θα δουλέψουμε μαζί τους για τη, κάποια εργαστήρια στη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου για τα παιδιά γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ε, δομές κατάλληλες για να μπορέσουμε να διοργανώσουμε ε, τις ημέρες τους γιατί σχολεία δεν υπάρχουν και οι οικογένειες ε, θέλουν πολύ να προσπαθήσουν να, να αποκαταστήσουν την κανονικότητα του κοινωνικού ιστού. για να μπορέσουν να ζήσουν κάποιες θετικές εμπειρίες Πιστεύω πως οι νέοι, ε, τα παιδιά του Σώματος Ελεγγύης μπορούν ακόμα να προσφέρουν τη σημαντική του συμβολή για να βοηθήσουμε τον κόσμο να συνεχίσει και να προσπαθεί με την επιλογή των φρικτών αυτών σεισμών δηλαδή την προσπάθεια να μείνουμε στην πόλη μας. Τα παιδιά λοιπόν του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μας έκαναν να σκεφτούν ε, να σκεφτούμε και να καταλάβουμε πως δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί από πολύ μακριά πήραμε πολύ στοργή και ε, μας έκαναν και μας πρόσφεραν υπηρεσίες που μας έδειξαν ότι μπορούμε να υπάρχουν και άλλες πραγματικότητες ε, ακόμα και σε μια πόλη που χτυπήθηκε τόσο πολύ σκληρά από το σεισμό. Χάρη σε αυτό το μεγάλη αγάπη και αλληλεγγύη που ε, μπόρεσαν να μας προσφέρουν ε, αυτά τα παιδιά. Αυτή είναι η ελπίδα να μπορέσουν ακόμα να μας βοηθήσουν γιατί σήμερα ζούμε την πιο δύσκολη φάση γιατί είχαμε Τις μέρες αμέσως μετά, όταν έφτασαν πρώτη φορά τα παιδιά, είχαμε μια ανταπόκριση συγκινησιακή. Ε, Θελήσαμε να δείξουμε δηλαδή ότι θα τα καταφέρουμε να μείνουμε στην πόλη μας. Σήμερα ε, χρειαζόμαστε συγκεκριμένες απαντήσεις ε, και να ανοικοδομήσουμε. Όχι απαραίτητα όμως να ξαναφτιάξουμε γιατί μπορεί κάποιοι να επιλέγουν να μείνουν στο ίδιο μέρος αλλά πέρα από τα σπίτια πρέπει να υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα δηλαδή σχολεία, να κάνουν τα παιδιά αγγλικά Τώρα τα, οι νέοι αυτοί τα κάνουν τα μαθήματα, να έχουν, παιδιά, να έχουν παιδικές χαρές οι ηλικιωμένοι μας, να έχουν την ανάγκη να έχουν κάποιον με τον οποίο να συνομιλούν. Τα παιδιά αυτά έχουν κάνει τα ψώνια των ηλικιωμένων, έχουν μπει στα σπίτια των σεισμόπληκτων, στα σπιτάκια των ηλικιωμένων και βοήθησαν σε όλες αυτές τις πτυχές. Όλα αυτά είναι υπηρεσίες που σε ένα μέρος που δεν πλήγει από το σεισμό είναι ίσως φυσιολογικά, σε εμά αυτές οι υπηρεσίες επειδή πρέπει να σκεφτούμε άλλα πράγματα πρώτα, δεν υπήρχαν πια και οι νέοι μας τα προσέφεραν. Ελπίζουμε λοιπόν να θα συνεχίσουν να είναι κοντά μας και να μας βοηθήσουν να επανέλθουμε στην κανονικότητα. And very last conclusion. Τελευταίο συμπέρασμα. Νομίζω ότι πραγματική πρόκληση στην επικοινωνία μας είναι να βγούμε από αυτή τη φούσκα γιατί είναι εύκολο να μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο πολύ στο ίδιο μήκο κύματο, όπως οι άλλοι θελοντές αλλά αν το μιλάμε σε κάποιον που δεν έχει σκεφτεί ποτέ τον αθλητισμό ως λύση πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε λοιπόν αυτή τη ε, φούσκα των στενών φίλων και γνωστών μας απάντηση θα θέλαμε να κάνουμε την αθλητισμό trendy της μόδας Κάποιοι ενδεχομένω να δουλεύουν ε, μόνο για χρήματα και αυτό μόνο να δέχονται. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να το κάνουμε μόδα, αν θέλετε. Θα μπορούσαμε να καλέσουμε λοιπόν κάποιους τέτοιους ε, influencers που κανονικά δουλεύουν μόνο επί χρήμαση για ένα τέτοιο project. Νομίζω ότι θα ήταν μια κατάσταση αμοιβαίου ωφέλους. Και αν κάποιοι άλλοι στη συνέχεια κάποια άλλη τέτοιοι σε δουν ότι αυτό βοηθάει η ιδέα της αλληλεγγύης. Φαντάζομαι ότι αυτό θα διαδοθεί ως μήνυμα και σε κοινότητες και ομάδες που δεν έχουν σκεφτεί εμ, τον εθελοντισμό. Ναι, καταλαβαίνετε. Χρειαζόμαστε κάποιον να μαγνητήσει. Έχετε κάνει κάτι στον τραντισμό. Όχι, όχι, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Ναι, θα σας ήταν πάρα πολύ ε, ευπρόσδεκτη στην Όρσια. Να ευχαριστήσω τον Νικόλα Αλεμάνο, τον Δήμαρχο της Όρσια, για την ε, πολύ συγκινητική του παρουσίαση, του Τζακ Άντερσον ε, από την οργανωσή και φυσικά την κυρία Καραπόσκα, η οποία μας έδωσε πολύ χρήσιμες σύμβουλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο πάνελ Thank you very much indeed. Now... Ευχαριστούμε πολύ. Αν πιστεύετε πως το ποδήλατο είναι καλό για την υγεία σας, είναι αλήθεια. Στην επόμενη ιστορία θα δούμε ότι μέσα από το ποδήλατο για την ποδηλασία μπορεί κανείς να ξεκινήσει μια λυσίδα αλληλεγγύης. Ας δούμε αυτό το βιντεάκι πρώτα. When biking meets charity and when boldness meets volunteering, here comes the Budapest Bike Mafia, introducing the charity team who ride the city day and night to help those in need.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 Another concrete example, Commissioner, this is... Ένα άλλο συγκεκριμένο παράδειγμα, Επίτροπε, είμαστε στην Ουγγαρία, στη Βουδαπέστη, μαζί με την ε, μαφία του ποδήλατου της Βουδαπέστης. Πολύ μου άρεσε αυτό το όνομα. Και εδώ θα βρούμε την Ιβλικο Τόρς που είναι εκπρόσωπος της ε, οργάνωσης ε, η μαφία του ποδήλατου της Βουδαπέστης.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 Η Ελιζαμπέτα Ρούζιτσις από την Κροατία που είσαι πρώην εθελόντρια ε, πέρασες πολύ χρόνο κάνοντας ποδήλατο στη Βουδαπέστη μου είπε χθε ότι ήταν η πόλη των ονείρων σου άφησε ακόμη και τη δουλειά σου για να μπει στο σώμα αλληλεγγύη. πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που θα μα την διηγηθεί σε λίγο και ο Ρόμπερτ Βάι, που δουλεύει σε ένα καταφύγιο στη Βουδαπέστη και παρέχεται εκεί βοήθεια στον κόσμο που το χρειάζεται και θα μα πει πώ αντιλαμβάνεται αισθάνονται τους εθελοντές ή ωφελούμενοι. Και τέλος δίπλα μου κάθεται ο Πάολο Ροντρίγε που πολύ ε, τον ξέρετε ως ε, Λετσίκο Πάολο που είναι blogger ε, με έδρα τη Γαλλία. Αν μπορείτε, θέλετε να μιλήσετε γαλλικά μπορείτε. Αν προτιμάτε τα αγγλικά είναι δικό σας θέμα. Ε, εμείς θέλουμε να μας πείτε πώς θα μπορούσαμε περισσότερο να διαδώσουμε αυτή την ωραία ιστορία. Ακούσαμε, είδαμε μόλις ένα βίντεο και θα, ακούσουμε, θα ξεκινήσουμε με την ελληνικό γιατί ήταν το δικό της, η δική της ιδέα. Πολύ ωραία η ανάμεξη ποδηλασίας με την αλληλεγγύη. Εσύ πώς ήρθες σε επαφή με το Σώμα Αλληλεγγύης και πώς σε βοήθησαν αυτό το, να προχωρήσει αυτό το project. Μάλιστα. Το, η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα ήταν κάτι νέο και ε, έφτασε με μένα στην οργάνωση γιατί είχα ήδη εμπειρία 10 ετών σε αυτό το project. Πριν από δύο χρόνια, το 2017, δημιούργησα το project αυτό και έκανα την αίτησή μου τον Οκτώβριο του 2017. Δύο μήνες αργότερα ήξερα ήδη πως εγκρίθηκε το project μου και έτσι προετοιμάσαμε μαζί με μια πολύ ωραία ομάδα του Budapest Bike Mafia το πρόγραμμά μας. Πέρσι το Μάρτιο έφτασε η Τόνια από τη Γερμανία, ε, μια συνάδελφο από την Φιλανδία και η Ελιζαμπέτα από την Κροατία. Το project σταμάτησε το περασμένο Δεκέμβριο. Μπορώ να σας πω πως ήταν μια φανταστική ιδέα που για όσους συμμετείχαμε γιατί, γιατί η μαφία του ποδήλατου ε, πήρε πολλά από αυτά τα τρία κορίτσια και όλες τις δυνατότητες που δίνει αυτό το πρόγραμμα σε μας. Τα κορίτσια έφτιαξαν το δικό τους πρόγραμμα στη διάρκεια των 8, 8 μηνών και μπορούμε να βασιστούμε σε αυτό το πρόγραμμα, μπορούμε να το βάλουμε στην εθελοντική μας δουλειά. Θα πρέπει να γνωρίζετε πως η μαφία του ποδηλάτου είναι μόνο εθελοντές. Έχουμε δηλαδή δουλειά και βοηθάμε στον ελεύθερο χρόνο μας. Επίση, γι' αυτό τον λόγο, τα τρία αυτά κορίτσια μας βοήθησαν πάρα πολύ. Η Ρόνια έφτιαξε το όνομα στο Βρετανικό Διεθνές Σχολείο που δουλεύει με τα παιδιά. Η Ελιζαμπέτα δημιούργησε ένα project σε ένα καταφύγιο αστέγων όπου ο κόσμος που ζει εκεί είχαν, είχε τη δυνατότητα να έρχεται μαζί της σε επαφή τακτικά και πιστεύω πως όλες αυτέ οι δυνατότητες έκαναν τη ζωή των αστέγων καλύτερη. Την έφεραν σε ένα διεθνές περιβάλλον και νομίζω αυτό ήταν πολύ καλή ιδέα. Να ακούσουμε τώρα την ε, ε, πρόταση πρόταση εγώ ήμουν online, είδα το project και ήξερα ότι εκεί θέλω να πάω. Ναι, εγώ δούλευα στην Κροατία, στο Ντουμπρόβνικ, ε, στη πόλη του Game of Thrones, δίπλα στην παραλία. Και ήταν ε, σαν μια ιστορία του ίντερνετ. Είχα καλή δουλειά, όλα ήταν τέλεια, αλλά κάτι μου έλειπε. Και υπήρχε αυτή η ανάγκη να είμαι και εγώ κομμάτι της κοινωνικής δουλειάς. Κάποια στιγμή λοιπόν άρχισα να ψάχνω στο ίντερνετ, έψαχνα ένα project ε, που να θέλω να συμμετέχω και είδα Budapest Bike Mafia, η μαφία του ποδήλατου της Βουδαπέστης και είπα πω πω τι είναι τούτο. Ε, ήρθα σε επαφή με την Ιόρντι και μετά από την αίτησή μου αποφάσισα να τα μαζέψω και να μετακομίσω στην Βουδαπέστη. Όταν έφτασα εκεί είδα ότι ήταν καλή απόφασή μου γιατί η μαφία του ποδήλατου για μένα είναι κάτι τελείως διαφορετικό κάνουν κάτι επιτόπου. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω καν. Δηλαδή προσπαθούν να εξισορροπήσουν τις καθημερινές τους δουλειές με την, τον εθελοντισμό. Και έχουν πολλά διαφορετικά project μέσα στο project. Είναι πολύ ενδιαφέρον λοιπόν. Ναι, είναι πράγματι. Πόσο καιρό πέρασες στη Βουδαπέστη, έξι μήνες. Έξι μήνες και βοηθούσες ε, λοιπόν τον κόσμο που ερχόταν και μιλούσε μαζί σου για τα προβλήματά του και δεν μιλάς ουγγρικά. Και δεν, πώς, είναι πολύ δύσκολη γλώσσα τα ουγγρικά. Πώς επικοινωνούσες. Εγώ είχα κάποιον ε, μεταφραστή, διαρμηνέα δηλαδή, που μιλάει ουγγρικά και αγγλικά. Και είναι πάντω εντυπωσιακό να είναι ένα κορίτσι από την Κροατία που ήταν έτοιμο να φύγει και να πάει να δουλέψει. Εγώ, δουλε... όταν δούλευα στο καταφύγιο ο κόσμος με έβλεπε με χαρά, προσπαθούσαν να μιλήσουν μαζί μου, κάποιοι ξέραν κάποιες λεξούλες κροατικά, είχε πλάκα. Μα έλεγε ε, ότι είχες μια φοβερή δουλειά σε Στην όμορφη πόλη, ε, την πόλη του Game of Thrones, αλλά προσπα... ήθελες να έχεις περισσότερο νόημα στη ζωή του. Το βρήκε, Ναι, ναι, βέβαια. Εγώ βρήκα τον εαυτό μου στη Βουδαπέστη. Και πώς το μετέφερες αυτό στην Κροατία? Ε, μα δεν πήγα ποτέ πίσω στην Κροατία. Συνέχισα να ζω στη Βουδαπέστη λίγους μήνες μετά. Μετά αποφάσισα να πάω στη Λουθουανία και από τη Λουθουανία στη Γερμανία. Τώρα δηλαδή είμαι στη Γερμανία, στη Στουκάρδη. Και τι κάνεις εκεί. Επισκέφτομαι τη μητέρα μου. Έκανα αίτηση σε ένα πανεπιστήμιο στο Άμστερνταμ. Οπότε είμαι πανταχού παρούσα. Μάλιστα, οπότε από την Βουδαπέστη ξεκίνησε μια μακρά πορεία που ελπίζουμε να συνεχίσει με επιτυχία. Να στραφώ στο Ρόμπερτ, όπω είπα, εσεί φροντίζει ένα καταφύγιο στη Βουδαπέστη όπου βοηθά ανθρώπου που το χρειάζονται, που δεν έχουν σπίτι, είναι άστεγοι. Πώς ε, εντάχθηκαν οι εθελοντές στο ε, καταφύγιο έπρεπε να γίνουν κάποια βήματα γιατί στην αρχή ακόμα και εγώ και οι συνάδελφοί μου ήμασταν μπερδεμένοι πώς και τι θα κάναμε τι θα έπρεπε να κάνουμε, αν θα έπρεπε να φοβηθούμε ή όχι. Περισσότεροι φοβούνται. Αλλά ήρθε η Ελίζαμπετ και μας κατέκτησε όλους. Ε, γιατί ε, και για μας αλλά και για τους ε, ε, ε άνθρωπους που έρχονται εκεί είχε πολύ στενή επαφή και ήταν κάθε μέρα εκεί στο καταφύγιο και αυτό φάνηκε σε μερικές μέρες μόλις γιατί αν στραφεί σε κάποιον είτε είναι άστεγος είτε όχι και του δώσεις όλη σου την προσοχή σε λίγα λεπτά μόνο υπάρχει αυτή η επαφή και η Ελιζαμπέτα αυτό το έκανε πάρα πολύ καλά γι' αυτό και ήμασταν ευτυχείς που ήταν εκεί στο καταφύγιο είχε καλές ιδέες καλές ερωτήσεις και μας έδωσε feedback. Εκείνη ήρθε λοιπόν όντως από άλλη χώρα. Τι είδους feedback σας έδωσε. Θα σας πω, εγώ δουλεύω δύο χρόνια στο καταφύγιο και είχε μια πιο φρέσκια άποψη για το πώς θα έπρεπε να βλέπουμε τους ανθρώπους αυτούς, δηλαδή να μην δίνουμε μόνο δουλειά του ποδαριού ή αν έχω χρόνο να προσπαθήσω να μιλήσω μαζί τους και να κάνω ό,τι μπορώ, αλλά όχι, εκείνη είχε άλλη στάση. Κάθε στιγμή ήταν πολύτιμη για εκείνη και της έδινε ε, και νέα και μαθήματα. Εμείς την περισσότερη μέρα είχαμε να κάνουμε με χαρτιά, αλλά μας έδειξε πως ο άνθρωπος είναι αυτός που έχει σημασία. Πάντοτε είναι καλή μια εξωτερική συμβουλή. Να ρωτήσω την Ελιζαμπέτα. Αυτή η εμπειρία σας έκανε να συνειδητοποιήσετε ότι είμαστε όλοι Ευρωπαίοι πολίτες και ότι οι γλώσσες, τα, τα σύνορα, τα γλωσσικά δεν έχουν τόση σημασία. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι αυτή η αίσθηση ε, του να θες να βοηθήσεις βασικά, να, να, να κάνεις ό,τι κάνεις με πάθος. Ναι, όντως. Στην αρχή είναι αρκετά... Ε, ε, φοβίζει ε, μάλλον αρκετά κάτι τέτοιο, αλλά δεν θα έπρεπε κανείς να φοβάται γιατί όταν πάει σε μια άλλη χώρα βλέπει πόσες πόρτες ανοίγουν, πόσες ευκαιρίες θα έχεις γιατί κοιτάξτε τώρα σήμερα είμαι εδώ στην Ευρωβουλή Δηλαδή, αν κάποιο μου έλεγε 8 μήνε πριν ότι θα ήμουν εδώ στο Εύρω στι Ρηξέλλε, θα έλεγα Τι λε τώρα, σαν χλαμάρε, ανοησίε. Αλλά να με. Η οικογένειά σα τι είπε, τι, ποια ήταν η αντίδραση όταν τους είπατε θα παρατήσω τη δουλειά μου ή θέλω να γίνω εθελόντρια. Το ήξεραν γιατί από πολύ μικρή ήμουνα έτσι. Δηλαδή πάντα πάω κάπου, δηλαδή παίρνω ε, ένα σακίδιο στο πλάτη και πάω. Σα καταλαβαίνω όμω. Όχι, δεν με καταλαβαίνω. Πολύ δύσκολο να το εξηγήσω στην οικογένειά μου. Αλλά ε, καθώ περνά καιρό, προσπαθούν να καταλάβουν περισσότερο. Καλό είναι που τουλάχιστον προσπαθούν να καταλάβουν. Μάλιστα. Ελιζαμπέτα ε, ε, ε, Ίντλη, συγγνώμη. Έχετε περισσότερους εθελοντές σήμερα στη Βουδαπέστη. Ναι, τώρα προετοιμάζω το νέο project και θα ζητήσω, θα κάνω την αίτησή μου τον Οκτώβριο γιατί έχουμε ένα τακτικό εταίρο. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν το πρώτο μας project και όπως σας είπα είμαστε όλοι εθελοντές και κάποιες φορές ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά χωρί καλή ομάδα δεν θα είχε καταστεί δυνατό να τα καταφέρουμε για 9 μήνε ε, σύνολο. Και επίσης ε, θα συνεχίσουμε την ε, μαφία του ποδήλατου γιατί βλέπουμε πολλές δυνατότητες για τους νέους, για την ένωσή μας αλλά και για τον κόσμο που το χρειάζεται και που ήδη μας έχουν γνωρίσει. Χωρί να πούμε σε όλες τις λεπτομέρειες, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για κάποια οργάνωση, κάποια ένωση να συνδεθεί με το σώμα Όχι, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο καθόλου. Όχι. Είναι πολύ εύκολο. Πολύ πολύ εύκολο. Και για κάποιο συμμετέχοντα πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν να μπει εκεί και να ε, καλύψεις όλα τα στοιχεία. Είναι πολύ εύκολο γιατί υπάρχει στήριξη στη χώρα σου αλλά και στη χώρα που πας. Άρα είναι πολύ εύκολο. Και για κάποιον δικαιούχο φαντάζομαι ότι εσείς με ανοιχτέ αγκάλες καλωσορίζετε τους ε, θελοντές και λέτε θέλουμε κι άλλους, θέλουμε να συνεχίσουμε. Ναι, είμαστε πάντα έτοιμοι. Γιατί έχουμε πολλές δωρεές, ε, έχουμε θελοντές. Ε, εμείς ε, το διασκεδάσαμε, εμείς το ε, διασκεδάσαμε που τον είχαμε κοντά μας. Η, η, η, η άστεγοι ένιωσαν πιο άνετα. Τα σύνορα δεν, δεν υπάρχουν. Ενωμένοι στην διαφορά μας. Αυτό είναι ο ορισμός. Επίτροπε, εσείς έχετε να μας πείτε κάτι για αυτή την ε, ιστορία. Ξέρατε για την μαφία της Βουδαπέστης. Ναι, ναι, έχω ακούσει πολλά για και το πρόγραμμα, αλλά ποτέ δεν τους είχα συναντήσει. Είναι μια μοναδική ευκαιρία και για μένα. Βεβαίως ε, πάλι έχει να κάνει αυτό με το πνεύμα, το ευρωπαϊκό πνεύμα της αλληλεγγύης και αυτό γιατί το επίπεδο του θελοντισμού στις κεντρικές χώρες ε, της Ευρώπης και μάλιστα στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης είναι χαμηλότερο. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες δηλαδή μπορεί να όντως να ζωγονήσουν το ενέστηση αυτή του συμμετοχής του πολίτη, του θελοντισμού και πραγματικά εκτιμώ τις προσπάθειές σας και τη συνεργασία σας γιατί είναι ε, μια ιδιαίτερη περίπτωση συνεργασίας, ένα νέο είδος. Ξέρω ότι και η Κροατία έχει έχει παράδοση και ιστορία σε αυτό, αλλά είναι ένα νέο είδος συνεργασίας γιατί υπογραμμίζει τη σημασία καινοτομία και στην εθελοντισμό. Γιατί υπάρχουν αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι τομείς, οι θεσμοί που κάνουν τη δουλειά την εθελοντική, αλλά με τον παραδοσιακό τρόπο και ξαφνικά κάποιος έρχεται και ναι, δίνει μια νέα πνοή. Με νέες καινοτόμε μεθόδους και αυτό είναι το ίδιο σημαντικό και για μας και για ολόκληρη την Ευρώπη. Και άλλη μια ερώτηση από το Twitter. Ποιε ήταν τα συμφέροντα και σε ό,τι αφορά τι χώρε εταίρου στο Ευρωπαϊκό Σώμα και έχουμε καθόλου πληροφορίε για το πόσοι συμμετείχαν το, σε ό,τι αφορά τις χώρες εταίρους. Το, το σχέδιο είναι ανοιχτό και σε αυτούς. Ναι. Και όπως είπα και προηγουμένως ε, από την Τουρκία έχουμε πάνω από 16.000 ε, αιτήσει και από την Ισλανδία, την Νορβηγία Δεν βλέπω άλλα κράτη-μέλη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Μακεδονία, Λίχτενστάιν. Μπορεί να έχατε λοιπόν κάποιους θεραντές από την Ισλανδία. Ναι. Θα θέλαμε πραγματικά να είναι πολυεθνικό το συγκείμενο. Γι' αυτό θα θέλαμε λοιπόν συμμετέχοντες από διάφορες χώρες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας να υπάρχουν ε, συμμετοχές από διάφορες χώρες. Φιλανδία, Γερμανία, Κροατία, είπατε. Πολύ ενδιαφέρουσες ε, συμμετοχές. Είναι πολύ καλό λοιπόν που υπάρχει αυτή η χημεία. Τώρα, να καλέσουμε τον Τσίκο πάλι στο να πάρει το λόγο. Ε, online influencer μας είπατε πώς μπορούμε να προωθήσουμε αυτή την πολύ ωραία ιστορία. Να είμαστε ειλικρινεί. Είναι πολύ καλή ω ιδέα και ενθαρρύνει πολύ κόσμο, ε, προσελκύει πολύ κόσμο, έχει πραγματικά μεγάλο βάθος ως ιστορία. Τώρα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε κόσμο και είναι λίγο λυπηρό να το θέτουμε έτσι, αλλά πραγματικά θα πρέπει πραγματικά να δώσουμε μια εικόνα. Να αναπτύξουμε αυτή την πλευρά, την πτυχή. Και γι' αυτό λοιπόν ε, τα social media είναι ένας βασικός τρόπος. Όταν μιλάτε για κοινωνικά μέσα, μιλάτε για το Instagram, ναι, ναι, ναι, δουλεύω στο Instagram. Ποια είναι λοιπόν η ιδέα αυτή που έχετε, ίσως αφορά αυτή την... Για να... Η συνταγή σας για να πετύχουμε πιο καλά αποτελέσματα. Χθες σας συζητούσαμε για το θέμα αυτό και ξέρω ότι είναι λίγο επιφανειακό να το συζητάμε αυτό τώρα αλλά έχουμε πολλά κομμάτια στο Instagram ιστορίες ε, feeds, χρώματα όλα αυτά θα πρέπει να τα κατανοήσουμε για να προσελκύσουμε την την νέα γενιά, την μελλοντική γενιά. Αν το πετύχουμε λοιπόν αυτό, θα ήθελα να έρθω σε επαφή με τους influencers στη Βουδαπέστη. Όχι ως θεατές. Θα μπορούσαμε να ε, κάνουμε ένα παράδειγμα, ένα πείραμα. Να πούμε καταρχάς ότι σε πρώτη φάση θα στείλουμε ένα ε, mail σε όλους τους ε, συμμετέχοντες στο Instagram, να προτείνουμε μία εμπειρία και να πω και κάτι λίγο λυπηρό, αλλά όλοι οι influencers είναι κενοί. Όλοι. ζητούμε κάποιο νόημα στη ε, ζωή μας και χρειαζόμαστε κάτι πιο βαθύ, για παράδειγμα όταν προτείνει κάτι, κανείς κάτι πιο ε, βαθύ σε έναν influencer θα ανταχθεί. Να προτείνουμε λοιπόν ότι έναν influencer να του δώσουμε ένα ποδήλατο να ερευνήσει, να, να εξερευνήσει μια πόλη, να κάνει ό,τι θέλει. Θα δημιουργηθεί έτσι μια τάση. Και γι' αυτό τους ονομάζουμε influencers, επηρεαστές, γιατί δημιουργούν καινούργιες επιρροές. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Δεν θέλετε λοιπόν ο influencer να είναι παρατηρητής, θέλετε να συμμετέχει. Ναι, βεβαίως. Να ζήσουν μια ημέρα... Ναι, θα πρέπει ότι ο, να ξέρουμε ότι ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ξέρει όταν κάτι είναι φτιαχτό και επίπλαστο. Χρειαζόμαστε λοιπόν, και αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, Το πρώτο λοιπόν θέμα είναι να δημιουργηθεί μια πραγματική ε, συνείδηση, όχι μόνο για την αλληλεγγύη, αλλά για την οικολογία, το φεμινισμό, να δημιουργηθούν λοιπόν νέες τάσεις για τους ε, και για την κοινωνία και με τους επηρεαστέ μπορούμε να φτάσουμε πιο μακριά και να έχουμε να επηρεάσουμε την ε, νέα γενιά. Μιλάτε για το Facebook, για παράδειγμα. Το Facebook, εδώ ποιο χρησιμοποιεί Facebook. Χρησιμοποιεί κανεί το Facebook. Ε, το Facebook είναι για του ε, γέρου. Εγώ σα τα λέω έξω από τα δόντια. Είναι λυπηρό, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Σε τέσσερα χρόνια μπορεί να έχουμε να έρθει ένα άνθρωπο και να μα πει Α, δεν τα χρησιμοποιούμε πλέον ούτε καν Instagram, γιατί ο κόσμο κινείται πολύ γρήγορα. Χρειαζόμαστε ένα νέο τρόπο να, για να επηρεάσουμε τους νέους. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα να συμμετέχουν οι influencers. Πείτε μας, σε ό,τι αφορά την ορατότητα, τι χρησιμοποιείτε σε αυτή τη φάση. Instagram, Facebook, έχουμε την ε, σελίδα, τη σελίδα μας, έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram. Είναι βασικά τοπικοί χρήστες ή έχετε πρόσβαση και στο, σε κόσμο εκτός ε, Ουγγαρίας. Όχι, έχουμε και την ιστοσελίδα μας και στα αγγλικά και μιας και είμαι και ο Διεθνής Σύνδεσμος της Βουδαπέστης. Έχουμε και mail, έχουμε και μηνύματα facebook. Και πρέπει να σας πω ότι είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε και μη Ούγγρους που κοιτούν ε, την, ιστοσελίδα μας. Έχετε και ωραία dessert, ε, ωραίες μπλούζες. Δεν ξέρω κατά πόσο τις πουλάτε και αυτές online. Ναι, έχουμε διάφορα Μάλιστα. Συνοψίζοντα λοιπόν, τι θα θέλετε να συμβεί, πώ θα θέλατε να εξελιχθούν τα επόμενα πέντε χρόνια για την ε, bike mafia κυρίως σε ό,τι αφορά και την ε, βοήθεια από πλευρά των εθελοντών. Ξέρω πολλές λεπτομέρειες για το σώμα αλληλεγγύης και είμαι βέβαιη δεν θα έχουμε μόνο ένα νέο, ένα νέο καινούργιο project. Θέλω να ανανεώσω την σφραγίδα ποιότητάς μας. Θα ήθελα να έχουμε και πιο πολλούς ε, του πιο σε πιο πολλούς αφαιρεντές. Όσοι δεν γνωρίζουν ε, τι σημαίνει αυτό, αυτή ακριβώ η σφραγίδα ποιότητα έχει να κάνει με τον αριθμό των εθελοντών που μπορεί να δεχτεί κανεί. Εγώ θα ήθελα να έχω όχι μόνο τρει αλλά δέκα εθελοντέ. Γιατί σήμερα έχουμε 13 διαφορετικά project και είμαι βέβαιη ότι θα υπάρχει ευκαιρία συμμετοχή σε όλα τα project της ε, Budapest by Mafia. Εσείς ε, από τη Στουτγκάρδη. Ελίζαμπεθ, πώ θέλετε να αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία στο μέλλον. Θέλω να κάνω κάτι στον τομέα της ε, κοινωνικής ε, ε, κοινωνική εργασία και έχω, θέλω να σπουδάσω στο Άμστερνταμ. Και θέλετε σε τελική ανάλυση να έχετε τη δική σας ΜΚΟ. Ναι, ελπίζω, ελπίζω. Στο μέλλον, όχι στην Κροατία. Α, μάλιστα. Όπου αλλού, αλλά όχι στην Κροατία. Όχι, όχι, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Κάπου στην Ευρώπη, κάπου στον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω όλους σας. Να ευχαριστήσω την Ήλντι, τον Ρόμπερτ, την Ελιζαμπέτα και τον Παόλο για την ε, συμβουλές που έδωσε. Μας ε, εμπνέεται και ελπίζω ότι θα μειωθούν και οι ανάγκες γιατί πραγματικά θα είναι πιο λίγοι αυτοί που θα βρίσκονται στο δρόμο. Και ελπίζω ότι με τα δικά σα τα project θα μπορέσετε να συνεχίσετε να βοηθάτε του άλλου, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο αυτό το project. Ευχαριστώ Well, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ήταν μεγάλη έμπνευση να ακούσουμε τα δύο αυτά παραδείγματα και να πω ότι πιστεύω ότι 15.000 ε, εθελοντές βρίσκονται σε αποστολές, μάλλον ε, συμμετείχαν σε αποστολές στην Ευρώπη. και αυτό το project είναι τόσο εικονικό όσο και το πρόγραμμα Erasmus. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο για τη δουλειά των εθελοντών αυτών και μου αρέσει αυτή η ιδέα του τριγώνου γιατί αυτό θεωρώ ότι καταστεί πάρα πολύ, καταστά πάρα πολύ ξεχωριστή την εμπειρία αυτή και θα ήθελα να, κάνουμε να βγάλουμε άλλη μια φωτογραφία να ζητήσω από όλους σας να μετακινηθείτε προς το κέντρο της αίθουσας αλλά να ευχαριστήσω καταρχάς όλους σας, να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας. Thank you Ah non, non, non, non, non, je vais, je vais pas le laisser là. So, Okay, so everyone, the idea is to move slightly towards the center of the hemicycle. Ελάτε προς το κέντρο του ημικυκλίου για όσους κάθεστε στις ε, μακρινές σειρές, ελάτε προς το κέντρο για να έρθουν να βγουν όλοι μέσα στη φωτογραφία. I would actually invite all the speakers to come forward. Όσοι μιλήσανε, ελάτε μπροστά. Μην εξταπηδάτε. Κάντε τον κύκλο.